εβδομάδα με ναι, θλίψη μάθαμε για τον θάνατο του Ντουάρ Φεράν, του συναδέλφου. Εξελέγει ευρωβουλευτής το 2014. Ήταν επικεφαλή τη αντιπροσωπείας στο ΙΕΝΕΦ του Εθνικού Μετώπου και επίσης ήταν μέλος Επιτροπής ε, Γεωργίας και ανάπτυξη της Υπέθρου και μέλος επίσης της Μικτής κοινοβουλευτική Επιτροπής για την Τουρκία. Ο κύριος ε, Φερό, μετά από μια μακρά ασθένεια, ε, ανεχώρησε και ήταν πάρα πολύ κριτικός όσον αφορά αυτή του την ασθένεια και επέδειξε πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Έχει αφήσει μία σύζυγο και πέντε μικρά παιδιά. Και είχα την ευκαιρία πέρσι, κατά την ε, αποστολή μας στην Ιταλία στους σεισμοπαθείς, έχουμε την ευκαιρία λίγο να συνεργαστούμε. Και ακόμη και αν είχα άλλο όραμα από εκείνη για την Ευρώπη και άλλες ε, ιδέες θυμάμαι ότι συμφωνήσαμε όσον αφορά ε, τις ε, πολιτικές του πεπιθήσεις και θέλει το, με το Κοινοβούλιο να εκφράσει τα θερμά συλληπιτήρια στην σύζυγό του, στα παιδιά του και σε όλους όσοι ήταν οικοί του σε όλη του τη ζωή και σήμερα πενθούν τον ε, θάνατό του. Προτείνω να τηρήσουμε ενός λεπτού σίγη. Merci. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κέγγι, έχετε το λόγο. Υπάρχει πρόβλημα με το μικρόφωνο της κυρίας Κιέγγι. Δοκιμάστε άλλο μικρόφωνο, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από το Ενεγύκλιο να σκεφτούμε ότι αν εδώ πέρα ε, ε, ε υπάρχει ε, ε φανατισμός όσον αφορά το χρώμα του δέρματος να σκεφτούμε ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα οποία έχουν σχέση με αντίληψη για νοτερότητα φιλετική και κάποιοι ε, εμπνέονται από κάποιους πολιτικούς που χρησιμοποιούν τη γλώσσα του μίσους. Θα πρέπει επομένως αυτό να το καταδικάσουμε όλοι ανεξάρτητα από το, από το χρώμα του δερματός μας. Grazie Ευχαριστούμε κυρία Κέγκε. Πρόκειται για αυτό το οποίο έγινε στην ε, Ματσεράτα. Αυτό το, οποίο είναι απαράδεκτο, αυτό το οποίο είναι απεχθές και όλοι μας καταδικάζουμε απερίφραστα και απόλυτα τα, τα πρακτικά έχουν εγκριθεί όσον αφορά